Cari colleghi, buongiorno a tutti. Eh, mi scuso. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση με την οποία ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Αλλά μπορώ να τα διαλογήσω. Ή, εν πάση περιπτώσει, να το εξηγήσω. Ναι, Ήμουν σε μια συνάντηση με τους πρόεδρους των υποεπιτροπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ασφάλεια και την άμυνα σε μια συνάντηση με τους 27 ε, πρέσβεις της Ένωσης και όπως πολύ καλά γνωρίζει ο φίλος, αν το επιτρέπει, πρώην πρέσβης ε, της Ιταλίας στην Καμπούλ, η εφράδια των πρέσβεων είναι γνωστή και χρειάστηκε να παραμείνω λίγο περισσότερο. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα να με δω ακριβώς τις τρεις. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω εκ μέρου όλων σας τον κύριο Σέκουι που είναι μαζί μας για πρώτη φορά σε μια ανακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τον συγχαίρουμε γιατί είναι ναι ειδικό απεσταλμένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Αφγανιστάν, αλλά και από τον Ιούνιο του 2009, πάνω κάτω δηλαδή τι ίδιε μέρε όπου όλοι μα εκλεγήκαμε στι χώρε μα. Έγινε επίσης και είπα το εκπρόσωπος της Ένωσης για το Πακιστάν. Αυτή η διπλή εντολή αντικατοπτρίζει στο άτομό του την περιπλοκότητα όλη αυτή τη υπόθεση και την ε, κρίσιμη φάση στην οποία διανύουν αυτοί, αυτές οι δύο χώρες. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και του είπα του εκπρόσωπου θα συνεσυχιστεί. Ο προκάτοχος του πρέσβη Σέκου, ο δόκτωρ Βεντρέλ, πέντε φορές είχε έρθει εδώ μαζί μας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της εντολής του. Και συνεχίζεται αυτή η σχέση συνεργασίας που όλοι ευχόμαστε να είναι καρποφόρα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Επιτροπή μας εδώ και καιρό παρακολουθεί το θέμα του Αφγανιστάν και όλα τα θέματα και τις ε, κρίσιμες ε, περιόδους που έχει περάσει όλη αυτή η περιοχή. Αυτή τη στιγμή ε, Ξέρουμε πως έχουμε το λεπτό ζήτημα των εκλογών. Ε, είναι μια χώρα η οποία είναι τελείως ε, νεόφυτη στη δημοκρατία και χρειάζεται να γίνει περισσότερη εμβάθυνση και εδραίωση. Ελπίζουμε λοιπόν πως θα είναι καρποφόρος ο διάλογος μεταξύ μας και ε, σίγουρα είναι Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα αυτά θα ακούσουμε, που θα ακούσουμε, να ρωτήσουμε ποιες είναι οι μελλοντικέ προπτικές της ε, κυβέρνησης του, Αφγανιστάν και σε σχέση με αυτό ποια θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας σε, αυτήν... σε αυτό το σενάριο, δηλαδή όσον μας αφορά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμμετοχή. Υπάρχει ακόμα ένα κρίσιμο σημείο που αφορά τον συντονισμό ανάμεσα στους διάφορους φορείς της διεθνούς κοινότητας. Υπάρχουν και αποκλήσεις που έχουν προκύψει πρόσφατα, το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε, να σταθούμε, ποιες θα ήταν οι προτάσεις του ή οι διευκρινήσεις που θα μπορούσε να μας προσφέρει στην Επιτροπή μας για αυτά τα θέματα. Οι συνάδελφοι σίγουρα θα θελήσουν να υποβάλουν ερωτήσεις ή να σχολιάσουν τα όσα θα ακούσουμε, αλλά σίγουρα θα αγγίξουν το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή και πιο συγκεκριμένα τους νόμους που εγκρίθηκαν και έπειτα κάπως αναθεωρήθηκαν, αλλά όχι σίγουρα με τον τρόπο που έχουμε εμεί συνηθίσει εδώ στις χώρες μας τα δικαιώματα της γυναίκας, περισσότερο από ότι αυτό του ανθρώπου γενικότερα. Επιτα υπάρχει δυνατότητα μιας εκλογικής μεταρρύθμισης εν ώψη των μελλοντικών προεδρικών εκλογών που θα γίνουν το 2010 και θα θέλαμε να γνωρίζουμε κάποια ίσως χρήσιμα στοιχεία για να κατανοήσουμε αυτή την εξέλιξη. Στη συνέχεια, η κατάσταση της, του εμπορίου ναρκωτικών. Υπάρχει μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα που περιέχει πολύ ανησυχητικές πτυχές. Και έλεγα στην αρχή πως ο πρέσβης Σέκουι συνδυάζει μια διπλή εντολή για τις ε, δύο χώρες, Αφγανιστάν και Πακιστάν, που από κοινού συμβάλλουν ε, στην κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη αυτή την περιοχή. Ποιε είναι οι πιθανότητε σταθερότητα ε, εκεί, ποιε είναι οι πιθανότητε οι δύο χώρε αυτέ να συνεργαστούν μεταξύ του. Και μια τελευταία παρατήρηση στα όσα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε αυτή την σύντομη εισήγηση που κάνω. Ποιο θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπο τη ιστορική διάσκεψη κορυφή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Πακιστάν που έγινε τον περασμένο Ιούνιο στι Βρυξέλλε. Αυτά και άλλα θέματα είναι αυτά τα οποία μας απασχολούν και στα οποία θέλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με χαρά δίνω το λόγο στον φίλο και μέγα συνεργάτη των ε, θεσμικών μας οργάνων, τον Έτορε Σέκουι. Σας ευχαριστώ. Ήρθα χθε το βράδυ επί τούτου από την Καμπούλ και θα επιστρέψω εκεί αμέσως μετά από την συνάντηση αυτή. Η κατάσταση είναι σίγουρα εξαιρετικά περίπλοκη αυτές τις μέρες στο Αφγανιστάν. Ακριβώς για να απαντήσω σε αυτή την ευγενική πρόσκληση και όπως και στην περίπτωση του προκατόχου μου ελπίζω ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Η τιμή που μου κάνατε να με έχετε εδώ σήμερα είναι γιατί είδα, σας είδα αγαπητέ Πρόεδρε, στο υψίπεδο μεταξύ Καμπούλ και Τζαλάλα Μπάντα σε πολύ επικίνδυνη περιοχή, ενώ εσείς διευθύνατε τις εργασίες για να κατασκευάσετε ε, μια γέφυρα. Επίσης να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο Προβέρα, αν μου το επιτρέπετε, γιατί είναι το άτομο χάρη στο οποίο κατά κάποιο τρόπο εγώ βρίσκομαι σήμερα στο Αφγανιστάν. Διότι όταν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιταλικής Γερουσίας, πριν από πέντε χρόνια, εμπιστεύθηκε έναν νέο που είχε την πρόθεση να πάει στο Αφγανιστάν και κατέστησε δυνατή αυτή την ε, αναχώρηση. Πρόεδρε Προβέρα, σας ε, θεωρώ, αν μου το επιτρέπετε, υπεύθυνο για τη σημερινή μου παρουσία εδώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι συνάδελφοί μου προετοίμασαν για μένα μια ε, ιδιαίτερα ε, εφράδη ομιλία, την οποία δεν πρόκειται να σας διαβάσω. Και αυτό διότι προτιμώ να σας κάνω μια πιο άμεση παρουσίαση για τις κατάστασης. Αν είχα διαβάσει αυτή την ομιλία, θα ξεκινούσα από την κατάσταση της ασφάλειας. Είναι γεγονός ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε αύξηση της ανασφάλειας στο Αφγανιστάν. Αν συγκρίνουμε την κατάσταση μεταξύ 2007 και 2009, οι περιοχές ανασφάλειας στο Αφγανιστάν έχουν αυξηθεί. Η ανταρσία στο Αφγανιστάν προσπαθεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του Αφγανιστάν, οι οποίες αυτή τη στιγμή θεωρούνται σχετικά πιο ασφαλείς. Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι η ματέωση που νιώθουν οι Αφγανοί ή τουλάχιστον κάποια κομμάτια της αφγανικής κοινωνίας, διότι δεν έχουν πραγματοθεί οι προσδοκίες τους. Θέτουν όλο και περισσότερο το ερώτημα κατά πόσο έχει βελτιωθεί η καθημερινή μου ζωή τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύπλοκο βέβαια το ερώτημα αυτό. Μετά από το 2001 οι προσδοκίες για βελτίωση της καθημερινής ζωής στο Αφγανιστάν ήταν έντονες. Το να ανοικοδομηθεί και να αποκατασταθεί μια χώρα μετά από 30 χρόνια πολέμου βέβαια δεν είναι απλό. Το άλλο πρόβλημα όμως, ο άλλος ιός αν θέλετε, και που έχει και χαρακτήρα παράδοξο, είναι η κόπωση των δωρητών. Η κόπωση των δωρητών από τις χώρες μας. Ενώ τα αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνουμε στο Αφγανιστάν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ικανοποιητικά. Αναφέρθηκατε τι εκλογέ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι ίσω το πιο καυτό θέμα αυτή τη στιγμή στη συζήτηση για το Αφγανιστάν. Η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εξ αρχή ιδιαίτερα σαφή σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία. Υποστηρίζουμε, <clears throat> είχαμε πει, την εκλογική διαδικασία. Δεν είμαστε εναντίον οποιοδήποτε υποψηφίου. Η εκλογική διαδικασία είχε φτάσει πια στο πέρας της και ένας δεύτερος γύρος, εάν είναι απαραίτητος, θα πρέπει να λάβει χώρα μέσα στον Οκτώβριο. Γιατί μετά τον Οκτώβριο, το χειμώνα, είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει η πολύπλοκη οργάνωση των εκλογών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτούς μας να συνεχιστεί η πολιτική αβεβαιότητα. Υπάρχει λοιπόν κόπωση των ίδιων των Αφγανών σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική διαδικασία. Είναι επίσης κεφαλαιόδες να εξασφαλίσουμε ότι η επίσημη εκλογική διαδικασία θα πρέπει να φτάσει στο πέρας της. Εμείς βασιζόμαστε σε δύο θεσμούς, την ανεξάρτητη Επιτροπή για τις εκλογές που αποτελείται από Αφγανούς και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι ένας ο πρώτος αφγανικός εκλογικός θεσμός μετά από 30 χρόνια και η ICC, η Διεθνής Επιτροπή, που έχει τέσσερα, τρία μέλη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και δύο Αφγανούς και οι οποίοι αυτή τη στιγμή εξετάζουν τη διαδικασία σε ορισμένα εκλογικά τμήματα και ελπίζουμε θα καταλήξουν σε αποτέλεσμα οι εργασίε του στο ταχύτερο δυνατό. Το επίσης σημαντικό ερώτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Το Αφγανιστάν χρειάζεται μια αξιόπιστη και δεσμευμένη να συνεχίσει η κυβέρνηση. χρειάζεται να υπάρξει ένα νέο συμβόλαιο μέσα εισαγωγικά μεταξύ της κυβέρνησης και των Αφγανών που να βασίζεται σε ένα πολιτικό μανιφέστο από την πλευρά του νικητή των εκλογών. Υπάρχει υποστήριξη για να γίνει μια διεθνής διάσκεψη στην Καμπούλ και η κυβέρνηση, νέα κυβέρνηση, <clears throat> χρειάζεται να καταδείξει ότι είναι υπεύθυνη, ότι είναι υπόλογη και ότι είναι προσιλωμένη στην δημοκρατική πορεία. Βέβαια, στο πλαίσιο αυτό έχουμε και καλά και άσχημα νέα. Υπάρχουν καταγγελίες για ατασταλίες και απάτες σε σχέση με την εκλογική διαδικασία. Και η Επιτροπή Εκλογικών Παραπώνων τα, τα εξετάζει όλα αυτά τα θέματα. Αλλά υπάρχουν και θετικά νέα, <clears throat> καταρχήν. Ήταν μια πάρα πολύ έντονη και ζωντανή εκλογική εκστρατεία. Η εστίαση της συζήτησης ήταν για τα εκλογικά προγράμματα και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των εκλογέων έγιναν παραδείγματο χάρη συζητήσεις μεταξύ των υποψηφίων. Στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Εκατομμύρια Αφγανών παρακολούθησαν αυτή τη συζήτηση και έθεσαν ερωτήματα, ζητούσαν απάντηση στα ερώτηματά τους επί τη βάση των εκλογικών προγραμμάτων για το ποια λύση θα έδιναν οι υποψήφοι στη χώρα. Ήταν επίσης ενθαρρυντικό ότι συμμετέχαν, συμμετείχαν όλες οι εθνοτικές ομάδες. Και οι δύο υποψήφοι, ο δόκτωρ Καζάη και ο Δ. Αβούλα, Αμπτουλά, πήραν ψήφους και σε περιοχές όπου η πλειοψηφία <clears throat> δεν ανήκει στη δική τους εθνοτική ομάδα. Θα πρέπει να θεωρήσουμε λοιπόν ότι αυτό αυτό το γεγονός ότι μπορέσαμε να οργανώσουμε εκλογές στο Αφγανιστάν ήταν μια επιτυχία. Φανταστείτε μια χώρα όπου πολλοί άνθρωποι σε πολλά χωριά δεν έχουν δει ένα μολύβι σε όλη τη ζωή. Πολύ περισσότερο μια κάλπη ή όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε 300 γαϊδάρους για να μεταφέρουν όλο το εκλογικό υλικό στα πιο απομακρυσμένα χωριά. Και υπήρξε και μια ομάδα Αμερικανών ε, κοινοβουλευτικών. Ένας από αυτούς, ο γερουσιαστής Φράνσις, μου είπε ότι αν σκεφτείτε ότι όταν εξελέγει εγώ την τελευταία φορά ήταν μικρή προσέλευση επειδή έβρεχε και δεν θέλανε να ψηφίσουν οι εκλογείς. Αν σκεφτείτε λοιπόν όλες τις απειλές που έχουν εκτοξευθεί από τους αντάρτες, του Ταλιμπάν, εναντίον των εκλογέων, υπήρξαν άτομα των οποίων κόπηκαν τα δάχτυλα, η μύτη από τους Ταλιμπάν. Νομίζω ότι ήδη το, η προσέλευση στις εκλογές καταδεικνύει ότι οι Αφγανοί θέλουν να είναι κύριοι της μοιρας τους. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, βασίζεται στο πρόβλημα της ασφάλειας. Ποια είναι η κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Η ασφάλεια είναι μια πολυεδρική έννοια. Υπάρχει η στρατιωτική πτυχή μέσα στο δόγμα του ΝΑΤΟ υπάρχουν διάφορες φάσεις του να εξασφαλίσει κανείς να διατηρήσει την ειρήνη και μετά να οικοδομήσει ένα νέο κράτος. Αλλά αν δεν μπορεί κανείς να διατηρήσει την ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομήσει. Υπάρχει λοιπόν αυτή η στρατιωτική διάσταση της ασφάλειας αλλά υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Μία από τις οποίες είναι η πτυχή της ανάπτυξης, η οικονομική πλευρά της ασφάλειας. Λέγαμε ότι πρέπει να κερδίσουμε και τις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Νομίζω πρέπει να κερδίσουμε και καρδιές και μυαλά και στομάχια. Γιατί χωρίς οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούμε πραγματικά να κερδίσουμε τον πληθυσμό και τις καρδιές και το μυαλό τους. Υπάρχει άλλη μια διάσταση όμως. Πιστεύω ότι η Ευρώπη <clears throat> πράττει πολλά στον τομέα αυτό και αυτή είναι η πλευρά η θεσμική της ασφάλειας. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει πολλές φορές στο Αφγανιστάν είναι ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο ιδίως σε τοπικό επίπεδο δεν είναι σε θέση να παράσχει τις βασικές υπηρεσίες στους πολίτες του. Τις βασικές υπηρεσίες που κάθε κράτος είναι υποχρεωμένο να τις παρέχει. Από την ασφάλεια μέχρι, μέχρι δικαιοσύνη, εκπαίδευση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σε όσες περιοχές λοιπόν μπορούν οι αντάρτες να ενισχύουν τη θέση τους γιατί δεν υπάρχει καμία παρουσία του κράτους. Σκεφτείτε το γεγονός ότι 60% των περιπτώσεων που θα πρέπει να έρθουν στα δικαστήρια, που έχουν να κάνουν με κτηματικές διαφορές. Στην Ήπεθρο υπάρχει η δυνατότητα είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό με χρήση βίας ή να πάνε ενώπιον του καδί, ενώπιον του δικαστή. Αν δεν υπάρχει όμως δικαστής, αν ο δικαστής είναι ανίκανος ή αν είναι διεφθαρμένος, τότε τα άτομα χάνουν τα δικαιώματά τους. Αποστερούνται τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και τότε οι Ταλιμπάν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν δικαιοσύνη και να εφαρμόσουν αποφάσεις που δεν προέρχονται από την επίσημη δικαιοσύνη. Το ίδιο συμβαίνει και για την παιδεία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πάρα πολλοί θεωρούν <clears throat> θεωρούνται ότι κατά κάποιο τρόπο είναι το εργατικό δυναμικό των ε, Ταλιμπάν. Άλλοι λένε 50, άλλοι 70% πηγαίνουν στις τάξεις των Ταλιμπάν γιατί δεν υπάρχει άλλος εργοδότης στο Αφγανιστάν. Δεν υπάρχουν οικονομικές ε, εναλλακτικές λύσεις. Παίρνουν περίπου 300 δολάρια το μήνα. Δεν υπάρχουν όμως άλλες ευκαιρίες απασχόλησης. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτό το θέμα το θεσμικό της θεσμικής διάστασης, σημαίνει ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε <clears throat> ότι ορισμένα σφάλματα δεν πρέπει να διαπράττονται γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργείται υποστήριξη για τους Ταλιμπάν. Πρέπει να προωθήσουμε το ταχύτερο δυνατόν τη δημιουργία μιας Ακαδημίας Δημόσιας Δίκησης. Η χώρα χρειάζεται περισσότερους τεχνοκράτες, περισσότερους δημόσιους υπάλληλους και ιδίως στο τοπικό επίπεδο. Εγώ τονίζω ότι η αφγανική κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια η ίδια να δημιουργήσει απαραίτητε τομέ και όχι μόνο στην Καμπούλ, αλλά και στις επαρχίες. Και η Ευρώπη κάνει πολλά πράγματα. Η EUPOL μετά από δύσκολη εκκίνηση έχει καταφέρει να επιτύχει πάρα πολλά πράγματα και να εδραιώσει το έργο της. Η EUPOL παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες. Βοηθάει τα Υπουργεία του Αφγανιστάν για την μεταρρύθμιση στις κρατικές δομές και ιδίως στη μεταρρύθμιση της αστυνομία. Και η αστυνομία είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στο θεσμικό τομέα σε ό,τι αφορά ιδίως την ασφάλεια. Επίσης, η U-POL συνεργάζεται με τους Αμερικανούς στα πλαίσια της CTCA, της αποστολής των Αμερικανών, που είναι υπεύθυνη για τη μεταρρύθμιση της αστυνομία. Ιδίως στον τομέα <clears throat> της δημιουργίας ένα, ενός φορέα της αστυνομίας για τις ποινικέ διώξεις, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο τη στιγμή που υπάρχει υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας. Χρειάζεται επίσης συλλογή πληροφοριών κτλ. Αλλά μέχρι πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε υπηρεσία συλλογής αστυνομικού χαρακτήρα πληροφοριών, το οποίο είναι κεφαλαιόδες σε όλες τις αστυνομίες. Επίσης, ο δεσμός μεταξύ αστυνομίας και δικαστικής εξουσίας είναι σημαντικό. Είναι σημαντικός. Θέλω να κάνω λοιπόν μία έκκληση προς εσάς. Η EU ακόμα έχει περιορισμένο προσωπικό σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, απαρτίζεται από περίπου 270 άτομα που είναι διεθνείς αστυνομικοί. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι <clears throat> σε τελική ανάλυση εξαρτάται από την ε, θέληση των κρατών μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν αστυνομικές δυνάμεις, εκπροσώπους των αστυνομικών δυνάμεων στο, Αφγανιστάν. Σας ζητώ λοιπόν τη βοήθειά σα να ενισχυθεί αυτή η αποστολή που είναι κέρια για την ασφάλεια του Αφγανιστάν. Κάτι άλλο το οποίο για μένα είναι κεφαλαίωδες. Η περιφερειακή διάσταση τη παρουσίας μας στο Αφγανιστάν. Πολλές φορές θεωρήσαμε ότι το Αφγανιστάν είναι ένα μια ενιαία αιστεία κρίσης. Δεν είναι αλήθεια. Θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα για να έχουμε μια περιφερειακή αντιμετώπιση όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σχέση Αφγανιστάν και Πακιστάν ή Αφγανιστάν με τις όμορες χώρες, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να σκεφτούμε την ευρύτερη περιοχή, όποιο είναι σε θέση να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη σταθερότητα του Αφγανιστάν στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να συμμετάσχει στις δραστηριότητες αυτές και πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων το Αφγανιστάν να γίνει ένα σταθερό κράτος που να έχει φιλικές σχέσεις σε όλους, αλλά πελάτης κανενός. Να είναι μια χώρα η οποία σταματά να εισάγει ασφάλεια και αρχίζει να εξάγει ασφάλεια. Υπάρχει ένα θέμα κύριε Πρόεδρε το οποίο δεν αναφέρατε. Η άποψή μου είναι ότι αυτό είναι το θέμα πάρα πολύ σημαντικό, είναι το θέμα της συμφιλίωσης. Αν μιλάμε ανοιχτά για το θέμα της ε, συμφιλίωσης με τους Ταλιμπάν, θέλω να σας προσφέρω τη δική μου άποψη για το θέμα αυτό. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι δεν μου αρέσει η έννοια συμφιλίωσης. Ούτε στα ντάρι, στην τοπική γλώσσα αυτή, αυτή η έννοια υπάρχει προτιμώ να χρησιμοποιήσω μια άλλη διατύπωση, που είναι η διατύπωση της συμπερίληψης. Συμπερίληψη σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Ότι πρέπει, το ερώτημα είναι αν πρέπει να έχουμε επαφή με αυτού οι οποίοι σήμερα αναφέρονται ω αντάρτες ή ως Ταλιμπάν. Η ω ταλιμπαν η απαντηση μου είναι ναι, αλλά με την προπόθεση ότι υπάρχουν ορισμένε κόκκινε γραμμέ που δεν θα τι διασχίσουμε. Καταρχήν πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ συμφιλίωσης και επανενσωμάτωσης. Η επανενσωμάτωση αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν κουραστεί να πολεμούν. Αυτούς που είναι το εργατικό δυναμικό των Ταλιμπάν, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, τα άτομα τα οποία δεν έχουν ιδεολογικούς λόγους, αλλά μόνο υλικούς λόγους να συνεργάζονται με τους Ταλιμπάν. Και αν δούμε τους Ταλιμπάν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους εντάσσεται κανείς στους ε, Ταλιμπάν. Είναι πάρα πολύ κα, κατακαιρματισμένος ο χώρος των Ταλιμπάν. Αυτό είναι ένα κέριο σημείο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε για να καταλάβουμε το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν έχει αυτό το χαρακτήρα κατακαιρματισμένης χώρας. Υπάρχουν αυτοί τους οποίους έχει διαβρώσει η Αλκαϊδα. Άλλοι τίνουν περισσότερο να δρουν επειδή νιώθουν ότι τους έχει αποστερήσει η κυβέρνηση, επειδή θεωρούν ότι οι φιλετικές τους ομάδες, οι φάρες τους έχουν τεθεί σε μειονεκτική θέση εναντί άλλων ομάδων. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι απλώς εγκληματίες. Οι οποίοι βρίσκουν ότι το κάτω είναι ο κοινό τους εχθρός. Είναι αυτοί οι οποίοι κρατούν μια καιροσκοπική στάση. Να συνταχθούν με την κυβέρνηση ή όχι. Ιδίως άμα η κυβέρνηση είναι αδύναμη. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έρχονται από στρατόπεδα, από καταβλισμούς προσφύγων και οι οποίοι έχουν αποκοπεί από τις αιστείες τους και από το κοινωνικό τους περίγυρο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος κατακαιρματισμός ακόμα και στις τάξεις των Ταλιμπάν. Τώρα για το θέμα της συμφιλίωσης. Νομίζω ότι όλα θα πρέπει να βασιστούν σε ορισμένες αρχές. Καταρχήν το σεβασμό του συντάγματος, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο ως σημείο αναφοράς. Γιατί στο Σύνταγμα έχουμε ορισμένε κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να τις περάσουμε. Καταρχήν έχουμε ένα καθεστώς συνταγματικής δημοκρατίας. Δεν μπορεί να είναι ένα Ισλαμικό Εμμυράτο. Το Σύνταγμα αναγνωρίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λοιπόν να υπάρξει παραβίαση αυτής της αρχής και οι γυναίκες να μην μπορούν να πάνε σχολείο. Το Σύνταγμα επίσης έχει σαν απαράγραπτη αρχή το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ούτε και αυτό μπορούμε να δεχτούμε να παραβιαστεί. Αν λοιπόν αυτή η διαδικασία, αν αυτή η πολιτική διαδικασία, η οποία βασίζεται στο Σύνταγμα, τη δέχονται ορισμένοι, είναι ανοιχτός ο χώρος ο συνταγματικός για αυτούς που την αποδέχονται και θέλουν να συμπεριληφθούν στην κοινωνία του Αφγανιστάν. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η συμφιλίωση πρέπει να γίνει μονάχα σε εθνοτική βάση, να αφορά μονάχα μια εθνοτική ομάδα. Θα πρέπει να δουν ότι πρέπει όλες οι ομάδες να συμμετέχουν. Θα πρέπει η διαδικασία να είναι αφγανική διαδικασία με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, αλλά μια αφγανική διαδικασία μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Με την προϋπόθεση συγχρόνως ότι η διαδικασία αυτή γίνεται αποδεκτή και από τις άλλες περιφερειακές δυνάμεις και τους περιφερειακούς παράγοντες. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. <clears throat> Νομίζω ότι η Ευρώπη ήδη κάνει πολλά. Νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερο. Καταρχήν, η Ευρώπη από το 2002 μέχρι σήμερα έχει δώσει πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ στο Αφγανιστάν. Και αυτό είναι μη στρατιωτικού χαρακτήρα υποστήριξη. Η Ευρώπη δρά σε σημαντικές περιοχές σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση, τη γεωργία, τη δημόσια υγεία κτλ. Έχουμε αναπτύξει μια αποστολή υγιού, όπως ανέφερα προηγουμένως, και ένας πρώην συναδελφός σας, ο Τζέιμορ Γιόγκ, ήταν επικεφαλής της ε, Επιτροπής Παρακολούθησης του ΟΗΕ, που ήταν μεγάλη σημασία όχι μόνο για να παρακολουθηθεί η διαδικασία προεδρικών εκλογών, αλλά και για να υπάρξει η προετοιμασία και της υποστήριξης σε ένα κύκλο εκλογικών διαδικασιών, γιατί πρέπει να ξεχάσουμε, όπως μας θύμισε ο πρόεδρος της Επιτροπής σας, ότι του χρόνου θα γίνουν κοινοβουλευτικές εκλογές και για πρώτη φορά εκλογή τοπικών συμβουλίων σε τοπικό επίπεδο που έχουν τεράστια σημασία γιατί είναι η πρώτη επαφή πολλών ανθρώπων με θεσμούς σε τοπικό επίπεδο. Όσο ο πρόεδρος και οι βουλευτές είναι στην Καμπούλ, τα τοπικά συμβούλια είναι αυτά τα οποία εκπροσωπούν τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο. Αυτά λοιπόν είναι η πρώτη γραμμή των αφγανικών θεσμών. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι όλες οι σημαντικές διασκέψεις για το Αφγανιστάν έχουν λάβει χώρα στην Ευρώπη. Στη Βόνη, στο Λονδίνο, Παρίσι, Χάγη, Ρώμη και υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και άλλες συνδιασκέψεις. Όλα αυτά έχουν μεγάλο νόημα, συγχρόνως όμως οι Αφγανοί κατανοούν τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Τι είναι όμως η Ευρώπη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε και η δική μου απάντηση είναι η Ευρώπη είναι μια περιοχή κοινού συστήματος και κοινών αξιών. Μεταξύ αυτών των αξιών είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι το λογοδοτήν από τις κυβερνήσεις, είναι η διαφάνεια. Αυτά ακριβώς τα οποία χρειάζονται οι Αφγανοί. Θέλω να προχωρήσω όμως και ένα βήμα περισσότερο και να πω ότι η ευρωπαϊκή οικοδόμηση βασίστηκε σε δύο βασικές έννοιες. Τον ιδεαλισμό αλλά και τον ρεαλισμό και βασίστηκε στην επικράτηση κοινών συμφερόντων <clears throat> και όχι των αμοιβαίων αντιπαλωτήτων. Αν το μεταφέρουμε αυτό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο Αφγανιστάν, σε μια χώρα όπου είναι δρεωμένη η καχυποψία μεταξύ των διαφόρων ομάδων, όπου όπου υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε οικονομικό επίπεδο που θα προκύψουν <clears throat> από μια συνεργασία, γιατί η ευρωπαϊκή οικοδόμηση βασίστηκε στην ενέργεια, στο άνθρακα και στο χάλιβα. Δεν μπορούμε να τα προσφέρουμε όλα <clears throat> στο Αφγανιστάν, μπορούμε όμως να προσφέρουμε την εμπειρία μας. Τι μπορεί να κάνει το Κοινοβουλίο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίδιος. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κρίνετε εσείς και θα ήθελα να τονίσω ότι εγώ προσωπικά πιστεύω στην κοινοβουλευτική διπλωματία. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία, διπλωματία είναι κρίσιμη και σε χώρες όπως ε, το Αφγανιστάν όπου είναι νεοσύστατοι θεσμοί και μπορούν τα κοινοβούλια να διαδραματίσουν πολύ πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Και μπορούν να εφαιρεθούν ε, από εσά οι καλύτερες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, ο πλούτος της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστείτε με την Αφγανική Βουλή, όσο γίνεται. Θα ήταν μεγάλη ενθάρρυνση κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό προσιλωμένοι. Γιατί είναι πολύ νεαρή χώρα το Αφγανιστάν. Το 60% του πληθυσμού ζει ε, μάλλον ε, δημογραφικά είναι κάτω της ηλικία των 30 ετών και αν συνεχίσουν έτσι οι δημογραφικοί δείκτες σε 15 χρόνια το 70 περίπου του πληθυσμού θα είναι ε, ηλικία κάτω των 20 ετών. Δηλαδή θα πρέπει να παραμείνουμε εκεί προσιλωμένοι για να μην χάσουμε ολόκληρη γενιά. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια κιόλας. Α, θα, τελειώνω. Πολύ σύντομα όμως, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ναι, ε, μήπως απαντώντας στις ερωτήσεις, αν θέλετε, σταματήσω εδώ και να τα πω τα υπόλοιπα μετά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβασή σας, Είστε τόσο πλήρη. Εγώ έκανα ερωτήσεις, ανέφερα θέματα και εσείς δώσατε απαντήσεις που θα παροτρύνουν τους συναδέλφους στη συζήτηση. Δύο σύντομες παρατηρήσεις καταρχήν. Επιτρέψτε μου προσωπικά να πω, ο πρέσβης ε, είχε την ευγένεια να θυμίσει μία σχετικά πρόσφατη περίσταση όπου συναντηθήκαμε στην Καμπούλ, όταν εκείνος ήταν ε, πρέσβης της, ε, της Ιταλίας, εγώ ήμουν δήμαρχος του Μιλάνου και μαζί κάναμε εργασίες για τη στήριξη μιας γέφυρας που είχε καταρρεύσει και γιατί ήμασταν εκεί, όχι γιατί ξαφνικά γίναμε ξυλουργοί, αλλά γιατί έφταναν από το Μιλάνο, γιατί το Μιλάνο είχε κάνει αυτό το δώρο στην πόλη της Καμπούλ, 49 λεωφορεία και 10 ε, συμπιεστές με τους οποίους διπλασιάσαμε τις δημόσιες ε, ε, μεταφορές της πόλης και στην ουσία αποκαταστήσαμε την ε, δυνατότητα περισυλλογής απορριμμάτων της πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Ε, όταν ε, μιλήσαμε για την κατάκτηση των καρδιών, πιστεύω πως αυτή η αποκατάσταση της γέφυρας είχε ένα νόημα ακόμα επίκαιρο. Σα ζητώ να είστε στα δύο λεπτά στι παρεμβάσει γιατί έχουμε λίγο χρόνο με τον πρέσβη και όπω φαντάζεστε λόγω του ενδιαφέροντος του θέματος έχω ήδη πολλούς συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Γι' αυτό σας ζητώ να σεβαστείτε αυτό τον χρονικό περιορισμό. Πρώτος θα πάρει το λόγο ο κύριος Μπέρμαν που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, με το Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πω Ολλανδικά καλύτερα, γιατί είναι η μητρική μου γλώσσα. Άκουσα τον κύριο Σέκουι και βλέπω ότι έχει προσωπικό θάρρος κάνει μια ανάλυση που με εντυπωσιάζει με σαφήνεια αλλά και συγκρατημένος και αυτό είναι και ο ρόλος σας εγώ θα περιοριστώ σε τρεις ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Μιλάτε για την ασφάλεια, για τη UPOL και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση της αφγανικής αστυνομίας της ίδιας για να βρει έναν τρόπο να ασφαλίζει την τάξη και την ασφάλεια. Έχω την εντύπωση ότι το δεν είναι μόνο πόσα επενδύει εκεί η Ευρώπη και σε χρήματα και σε προσωπικό, που είναι και αυτή σωστή ερώτηση, αλλά αυτή τη στιγμή τι εστί η αφγανική αστυνομία και τι θα πρέπει να είναι. Είναι η στρατιωτική προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών, η στρατιωτική μορφή αστυνομία τρόπον τεινά. Κάποιοι θερμοκέφαλοι ή ο αστυνομικός ας πούμε που ε, κυκλοφορεί ε, και περιπολεί σε μια συνοικία του Άμστερνταμ και σκέφτεται τι συνέπειες θα έχει αν συλλάβει κάποιον ας πούμε ή αν ε, τον επιπλήξει. Θα πρέπει να είναι μια αστυνομία που να σέβεται τον Αφγανό πολίτη και αν κάτι απέτυχε τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώς αυτό. Οι Αμερικανοί δηλαδή, πώς να το πω, που είχαν ε, τα χαρτιά στα χέρια τους και χάσαν αυτή την ευκαιρία τόσο γρήγορα. Λοιπόν, ποια αστυνομία βλέπετε εσείς να αναπτύσσετε και τι είδους αστυνομία. Ερώτηση δεύτερη. Τι εστί αφγανοποίηση του Αφγανιστάν. Αν θέλουμε σιγά σιγά να φύγουν ε, τα στρατεύματά μας και να έχουμε όλο και περισσότερη ανάπτυξη και ανοικοδόμηση, εσείς στην ανάλυση σας πώς φτάνετε στο να περάσει το Αφγανιστάν σε αφγανικά χέρια. Δηλαδή και ντόπιοι ηγέτες και τα Λιμπάν θα συμμετέχουν στη δίκηση της χώρας. Πώς το ορίζετε αυτό. Αυτά γιατί τελειώσαν τα δύο λεπτά μου και δεν μπορώ να κάνω άλλη ερώτηση. Ε, τα ξεπεράσατε και για τα 30 δεύτερα. Το λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος Κέλαμ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πολύ έμπειρη παρουσία σας ε, και είπατε ότι αν δεν μπορεί κανείς να προσφέρει κάποια ελπίδα δεν μπορεί να κερδίσει το νου και την καρδιά των ανθρώπων. Το ίδιο ισχύει όμως και για μας, για τις ε, χώρες ε, που έχουν συμμετάσχει στο Αφγανιστάν. Έχουμε 25 κράτη-μέλη που έχουν ε, άνδρες στο Αφγανιστάν. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική συνένεση. Ως εκ τούτου ε, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ υψηλό και ουσιαστικό και πολιτικά και οικονομικά. Αλλά η ελπίδα αρχίζει να αποδεικνύεται φρούδα και στην ε, Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε την άποψή σας για εναλλακτικές λύσεις στην ε, παρούσα κατάσταση. Φαίνεται ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι ο κύριος ε, Καρζάη τελικά είναι ο νικητής των εκλογών παρά τις ε, αμφισβητήσεις. Όμως η βιώσιμη δημοκρατία βασίζεται σε αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις και ρωτώ υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στον κύριο Καρζάη ίσως, ο κύριος Αμπτουλάχ, κάποιοι άλλοι. Πριν από 25 χρόνια οι άνθρωποι έλεγαν πρέπει να στηρίξουμε τον Κορμπατσόφ γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εμφανίστηκε τότε ο Γέλτσιν και είπανε το Γέλτσιν με κάθε τίμημα γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτών. Στη σημερινή έκδοση του Φίγκαρο ο πρώην επικεφαλής της ε, ΑΕΠ του Πακιστάν λέει ότι ο Μουλαχομάρ και ο κύριος ε, Καρζάι έρχονται από την ίδια πόλη και από την ίδια φυλή. Ως εκ τούτου, πιο κοντά δεν μπορούν να έρθουν. Και κάτι άλλο. Ε, εκταμεύσαμε πολλά χρήματα για την ε, επιστροφή των προσφύγων. Υπάρχει κάποια διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Αρλάκη έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Σέκουι, σίγουρα μπορούμε να ακούσουμε την έκκλησή σας για ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στο Αφγανιστάν και εκτίμησε ιδιαίτερα το θετικό σας πνεύμα σε σχέση με αυτά που πρέπει να γίνουν και τα ε, αποτελέσματα που θα πρέπει να επιτευχθούν, καθώς και την ε, ειλικρίνειά σας για τη δυσκολία να εργάζεται κανείς σε μια χώρα από τις πιο καταστραμμένες σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις, σας παρακαλώ, στο μέτρο του δυνατού να μου απαντήσετε, ίσω όχι με το 100% του τι σκέφτεστε, αλλά εν πάση περιπτώσει να μα επιτρέψετε να καταλάβουμε τι πιστεύετε. Είναι κάπω δύσκολες οι ερωτήσεις. Το πρώτο, ε, το θέμα του partnership. Νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα στο Αφγανιστάν. Με ποιο είδος κυβέρνησης ποιο είδος ε, προσωπικότητων με τη δική του συμμετοχή όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στο κοινοβούλιο και στην ε, περιφερειακή δίκηση τι πιθανότητες έχουμε να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν εναλλακτικέ, διότι από την ε, πολιτική μου σταδιοδρομία ξέρω ότι εναλλακτικέ πολιτικές υπάρχουν πάντοτε. Υπάρχουν ιδέες για το τι θα πρέπει να γίνει χωρίς τον Καρζάη και με κάποια άλλο είδος ε, συμμαχίας. Δεύτερη ερώτηση, το θέμα των ναρκωτικών για την οποία, το οποίο δεν μιλήσατε και το θέμα του crop elimination της ε, εξάλληψης αυτών των καλλιεργιών και των εναλλακτικών στην ε, οικονομία του οποίου. Ποιες είναι οι δυνατότητες της Ευρώπης και τον είπα. Ευχαριστούμε, ανακτήσαμε κάπως την καθυστέρηση, ότι ο λόγο έχει ο κύριος Αουτάλα. Κυρία, Κυρία συγγνώμη. I was listening to the Finnish interpretation, but they didn't mention my name. Συγγνώμη, άκουγα την φιλανδική μετάφραση, αλλά δεν μου ανέφεραν το όνομά μου. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Πιστεύω πως πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για το πολύ δύσκολο έργο το οποίο έχετε αναλάβει εξ ονόματός μας. Στην Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κοινοβουλίου πρόσφατα είχαμε ομιλητές από το Αφγανιστάν που ήταν ε, ε, πολύ ενημερωτικοί με όσα μας είπαν. Θα ήθελα να σας ζητήσω κάποια σχόλια για τα όσα ακούσαμε. Για παράδειγμα, είχαμε έναν ομιλητή από το Human Rights Watch, ε, την κυρία Rachel Reed από την Καμπούλ, και που είπε ότι ανησυχούν ακούσει ιδιαίτερα για τις πιθανές επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον προτινόμενο διάλογο με τους Ταλιμπάν και θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε. Επίσης ακούσαμε από το δίκτυο αναλυτών για το Αφγανιστάν που βασίζεται εδώ στην Ευρώπη αμφέβαλαν αν η εντολή για τις εκλογές για μια επιτροπή ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να αντισταθούν σε πολιτικές πιέσεις από τους ηθήνοντες της κυβέρνησης και την χειραγώγηση από πλευρά τους και γι' αυτό θέλω να ξέρω τι πιστεύετε και έπειτα εξετάζοντα κάποιε δυνατότητε σταθεροποίηση τη κατάσταση, ενώ βελτιώνεται η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ταυτόχρονα η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αστυνομία θα μπορούσε ίσως να προσέξει περισσότερο την, εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα της γυναίκας, ούτως ώστε να διαδοθούν αυτές οι αξίες τις οποίες θέλουμε να διαδώσουμε στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Το λόγο έχει η συνάδελφος Λέζινγκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την εκτενή σας παρουσίαση. Έχουν προκύψει και μερικά ερωτήματα για μένα και θα ήθελα να συνεχίσω από τον συνάδελφο που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας για το Αφγανιστάν, τον κύριο Μπέρμαν. Και ρωτώ, ε, ποιο είναι το μέλλον της αφγανικής αστυνομίας. Ήδη έχουμε ασχοληθεί στην Επιτροπή Ασφάλειας της ΣΕΝΤΕ και βλέπω ότι πολλοί από τις U-Poll είναι Γάλλοι χωροφύλακες ή Ιταλοί ε, από ε, που είναι παραστρατιωτικές ενώσεις αστυνομίας. Αυτό είναι πραγματικά άραγε πρότυπο για την Αφγανική αστυνομία. Δεν νομίζω ότι θα ήταν βήμα αυτό προς μια δημοκρατική εξέλιξη και μια πολιτική αστυνομία, μη στρατιωτική δηλαδή. Καμία σχέση δεν έχει με αυτά που εμείς στην Ευρώπη εκλαμβάνουμε ως αστυνομία, ούτε με τις δικές μας ευρωπαϊκές αξίες. Επίσης ρώτησε ο κύριος Μπέρμαν τι γίνεται με την αφγανοποίηση του πολέμου. Και εγώ ανησυχώ πολύ εκεί για τις εξελίξεις στη χώρα. Γιατί αν δούμε τι κράτος έχουμε τώρα στο Αφγανιστάν, η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη συνεργασία με εγκληματίες πολέμου και έχει πολύ χαμηλή ε, δημοτικότητα και στήριξη από τον πληθυσμό. Και ε, με ένα στρατό πάνωπλο, πανάκριβο, κοστίζει περισσότερα ε, ο εξοπλισμός από τον αφγανικό προϋπολογισμό της χώρας ολόκληρης. Πώς είναι λοιπόν Ε, να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Τι επιρροή έχουμε εμεί εκεί κύριε Πρέσβη στι ευρωπαϊκέ αποστολέ τη UPOL, Ευχαριστώ. ευχαριστώ κυρία Λέζινγκ. Το λόγο έχει ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Τρεις ερωτήσεις έχω. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στα σχετικά θετικά ε, σημεία της Ευρωπαϊκής Αποστολής που αναφέρατε κι εσείς. Και σας ρωτώ, κατά την άποψή σας, ποιο είναι το πιο θετικό στοιχείο που διαπιστώνετε εκεί. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόοδος για σας. Γιατί μιλήσατε για μαζική παρουσία της Ευρώπης εκεί και ότι έχουν ήδη γίνει πολλά. Ε, το καλύτερο από όλα αυτά που έχουν γίνει ποιο είναι. Ερώτηση δεύτερη. Σχέση Γιούπολ και ΝΑΤΟ. Μπορείτε να μας πείτε σας παρακαλώ ποια είναι τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας εκεί. Και αν υπάρχουν σημεία τριβής και δυσκολίες. Ε, και τέλος, αυτή είναι η τρίτη μου ερώτηση. Κάνετε μία διάσταση, μία διαφοροποίηση ανάμεσα στη συμφιλίωση και ε, την ένταξη ο πρόεδρος Καρζάη μιλάει για συμφιλίωση. Τώρα εσείς έρχεται να διαφωνήσετε με τον πρόεδρο Καρζάη. Είναι απλή η απόχρωση αυτή. Ευχαριστώ. Il primo round di interventi per due minuti l'onorevole Obiol. Και τώρα ο κύριος Ομπιόλ. Για δύο λεπτά. Είπατε ότι όταν αναλάβατε τα τόσα δύσκολα καθήκοντά σας, ε, το πιο δύσκολο εγχείρημα και αυτό που είχατε να αντιμετωπίσετε είναι να επικοινωνείτε με τις ε, Βρυξέλλες, με ε, τις φυλές των Βρυξελών. Σήμερα το έχετε καταφέρει. Είναι η 8η επέτειος της έναρξης σήμερα ε, των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και ενισχύεται η συζήτηση για το τι θα πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα χρειάζεται συνοχή και αυτό είναι απόλυτα σαφές ότι αποτελεί ε, προτεραιότητα. Μπορούμε να διαφέρουμε σε ερμηνείες μας, αλλά η πρόγνωση είναι ίδια, ότι η παρουσία η διεθνής στο Αφγανιστάν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα και θα παραμείνει σε παρατεταμένη περίοδο εκεί και σε αυτή την περίοδο θα πρέπει να χαράξουμε και ε, τις προτεραιότητές μας και πώς τις παρουσιάζουμε αυτές τις προτεραιότητες εκεί. Συμφωνώ πάρα πολύ ε, όταν λέτε ότι θα πρέπει να κερδίσουμε και το νου και την καρδιά αλλά και το στομάχι, ξέρετε. Εντάξει ο νους και η καρδιά, το στομάχι τι γίνεται. Ε, θα υπάρχει μια προτεραιότητα εκεί λοιπόν για το νου και την καρδιά, αλλά και μια ευθύνη για τα υπόλοιπα. Αυτά πολύ ωραία ορίζονται από την πρώην Πρωθυπουργό της ε, Νορβηγίας, Γκρό Χάρλεμ ε, που έλεγε το πιο σημαντικό είναι να ε, βελτιωθεί η ζωή των Αφγανών. Η Νορβηγία είναι στην πρώτη γραμμή ε, τη ευζοία και τη ευημερία. και τελευταίο είναι το Αφγανιστάν και ο Νίγηρα ως τόπος για να ζει κανεί. Και σας ερωτώ, και, ε, τι λέτε κι εσείς, γιατί ε, στις δημοσκοπήσεις όλος ο κόσμος του Αφγανιστάν αναφέρεται ως προβλήματα στην τροφή και στην υγεία του. Οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες ποιες είναι για να βελτιωθεί η ολέθρια κατάσταση της δημόσιας υγείας στη χώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Ομπιόλς. Ας αφήσουμε τον πρέσβη Σέκουι να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Για το θέμα της ε, αστυνομίας και της ασφάλειας υπάρχει μια έκφραση. Ε, σιωπηλό, σιωπηρό τσουνάμι. Αυτή χρησιμοποιείται στο Αφγανιστάν. Αυτό αναφέρεται στο γεγονός ότι καθημερινά, κατά μέσο όρο, 5-6 αστυνομικοί σκοτώνονται. Γιατί είναι σιωπηρό το τσουνάμι, γιατί κανείς δεν μιλάει γι' αυτό που συμβαίνει ή σχεδόν κανείς. Γιατί αν έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε στον ε, Guardian πριν από δύο μέρες υπήρξε μια διαρροή ε, μια δική μου έκθεσης όπου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω πως αυτή τη στιγμή, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται και η δυνατότητα να ε, περιορίζονται μέσω πολύ δυνατής αστυνομίας ώστε να είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε γιατί αυτό που πραγματικά είναι καταστροφικό για το Αφγανιστάν είναι όταν μια περιοχή καθαρίζεται και μετά δεν υπάρχει κανείς για να την κρατήσει. Μόλις φύγει η ασφάλεια επιστρέφουν οι Ταλιμπάν. Και ψυχολογικά είναι καταστροφικό αυτό. Αλλά είναι σαφές και αυτό είναι το όραμά μας ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα είδος ε, αστυνομία που πραγματικά θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική και να συνεργάζεται αποτελεσματικά και με το δικαστικό σώμα. Γιατί δεν μπορεί να κρίνει κανέναν αν ε, η αστυνομία δεν συλλαμβάνει κανέναν και τούμπαλιν. Αυτό που χρειάζεται να θεσπιστεί ακριβώ είναι και η εμπιστοσύνη για το ποιο αντιπροσωπεύει την ασφάλεια στην πόλη, για παράδειγμα. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, για ξέχασα να τον αναφέρει, είναι λάθος μου, αυτό που κάνει η αστυνομία είναι ότι αντιμετωπίζει ένα άλλο πρόβλημα που είναι η διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον νέο Υπουργό, βάση περιπτώσει, όχι και τόσο νέο, αλλά νέο, βάση περιπτώσει, αρχηγό, ε, Υπουργό μάλλον εσωτερικών, εάν αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαφθοράς στην αστυνομία και χρησιμοποιώ τα δικά του λόγια, τότε θα είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διαφθοράς. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομία ακριβώς αυτό προσπαθεί να κάνει. Για το θέμα της της ευγανοποίησης. Ευγανοποίηση τι σημαίνει. είναι η ανάθεση κάποιων δραστηριοτήτων στους Αφγανούς και κυρίως και πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Η πραγματική εφαρμογή μιας έννοιας, μιας ιδέας που είναι η κοινή, η λογοδοσία, αμοιβαία λογοδοσία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τη στιγμή που πραγματικά αποδοθούν οι διάφορες λειτουργίες ε, στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι κάτι το οποίο επαναλήφθηκε και στην Χάγη, στη διάσκεψη της Χάγης ότι δηλαδή αυξάνεται η διοχέτευση των ξένων κονδυλίων μέσω του προϋπολογισμού ε, προς τον ε, προϋπολογισμό του Αφγανιστάν. Αυτό θα πει αυγανοποίηση, αλλά τι σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιεί σωστά αυτά τα κονδύλια. Αυτή είναι η αμοιβαία λογοδοσία και αυτό ε, θα έτεινα να πιστεύω ότι αν δουλεύαμε προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις θα γινόταν σημαντικά βήματα μπροστά. Να σας πω μόνο ότι Κάποιες φορές τείνουμε να μιλάμε για στρατηγική εξόδου. Η αυγανοποίηση ίδια είναι μια στρατηγική, αλλά εγώ προτιμώ να την αποκαλώ μεταβατική. Μάλλον στρατηγική μετάβασης. Μετάβασης προς μια φάση όπου θα πρέπει να παραμένουμε βέβαια για μεγάλο χρόνο, αλλά οι βασικές δραστηριότητε τη χρηστή λειτουργία ενός κράτου συμπεριλαμβανομένη τη ασφάλεια θα είναι στα χέρια των Αφγανών. Πιθανές εναλλακτικέ στον Καρζάη. Ειλικρινά, από, από την αρχή έχω ερωτηθεί αυτό το, την ερώτηση και απαντώντας ανέκαθεν έλεγα το ίδιο πράγμα. τελικά οι Αφγανοί θα πρέπει να αποφασίσουν. Μπορούν να το κάνουν και θα πρέπει να αποφασίσουν. Και αυτό έτσι ώστε ο ηγέτης τους να είναι αξιόπιστος στα ίδια τους τα μάτια. Θα πρέπει μόνο τους να διαλέξουν τον ηγέτη τους. Νομίζω πως η καλύτερη εναλλακτική λύση είναι αυτή που οι Αφγανοί θα επιλέξουν οι ίδιοι για το θέμα των ε, προσφύγων. Και θα ήθελα καταρχήν να κάνω μια διευκρίνηση. Ο Καρζάη και ο Μουλά Ομάρ δεν ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο. Ο Καρζάη είναι μουλ, μου... Ανήκει σε άλλη φυλή από τον Μουλά Ομάρ. Μπας περιπτώσει, Υπάρχουν διάφορε φυλέ και σόγια από τα οποία προέρχονται. Εν πάση περιπτώσει, τα περιπλέξω. Είναι ήδη πολύ μπερδεμένα. Και για του πρόσφυγες είναι και αυτό θέμα κλειδί. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα των... της προέλευσης και νομίζω πως οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν πολύ γενναιόδορες σε αυτό. Το Αφγανιστάν ε, έχει στερηθεί εδώ και χρόνια των καλύτερων ανθρώπων τις καλύτερες ενέργειες που θα μπορούσε να έχει. Υπολογίζουμε, για παράδειγμα, ότι από 100.000 μέχρι 1 εκατομμύριο άνθρωποι, 900.000 μέχρι 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν γιατί ακριβώς βρίσκονταν εκτός της χώρας. Και θίγεται ένα θέμα κλειδί. Είμαι ευγνώμων για τα ερωτήματά σας και αντίθετα από τα όσα λέγονται, δεν είναι όλοι οι πρέσβεις ε, άνθρωποι που στέλνουν στο εξωτερικό ε, για να λένε ψέματα για τη χώρα τους. Εγώ εξάλλου έχω 27 χώρες που αντιπροσωπεύω. Πέρα από τα αστεία τώρα να σας πω το εξή. Η έννοια την οποία εσείς εκφράσατε ακριβώς είναι το θέμα επί του οποίου συζητάμε. Ε, δηλαδή είναι η επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα των εκλογών. Η διεθνής κοινότητα, θα πρέπει να πω και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκάθαρα, εξέφρασε μια ε, θέση η οποία πολύ σοβαρά λαμβάνεται υπόψη από όλου του Αφγανού πολιτικού. Ότι δηλαδή η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση που είναι στραμμένη προ το μέλλον και πολύ λιγότερο προ το παρελθόν. Και πέρα από το σύνθημα θα πρέπει να δούμε ότι η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στα πράγματα είναι εκείνη που εδώ και 4-5 χρόνια είναι η μόνη που έχει υπουργού ικανούς, ικανούς και επαγγελματίες. Αυτό λοιπόν που περιμένουμε να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών είναι οι υπουργοί που έχουν αποδείξει την αφοσίωσή τους στον επαγγελματισμό τους να συνεχίσουν να αποτελούν τμήμα του νέου πολιτικού συστήματος που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Και ο αριθμός τους μπορεί και να αυξηθεί. Επ' αυτού ε, είμαι αρκετά αισιόδοξο. Για το θέμα των ναρκωτικών. Δεν το ανέφερα επίτηδες. Θελημένα γιατί φαντάστηκα ότι θα μου κάνατε σχετική ερώτηση. Το θέμα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Γιατί αν δει κανεί και τα οικονομικά στοιχεία, δεν είναι μονάχα ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο εναλλακτικέ καλλιέργειε. Οι εναλλακτικέ καλλιέργειε, όπω ξέρετε και εσεί καλύτερα από μένα, είναι βέβαια πολύ σημαντικέ. Αυτό που λείπει είναι η διασφάλιση τη πρόσβαση στην αγορά αυτών των εναλλακτικών καλλιεργειών. Και γι' αυτό έχουν γίνει βήματα ε, μπροστά. Μπορούμε να μιλήσουμε, α πούμε, για την καλλιέργεια ελαιό, ελαιόδεντρων. Είμαστε πεπισμένοι ωστόσο πως η νέα κυβέρνηση μπορεί ε, να δεσμευτεί γι' αυτό και μπορεί ε, να δείξει και τα υπόλοιπα τους υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ε, πολλαπλασιάζονται δύο φαινόμενα. Από την μία έχουμε μία εγκληματικότητα η οποία καθοδηγείται από τους ίδιους παραγωγούς, είναι επιθετική και πολύ ισχυρή και είναι και υπερεθνική. Και το άλλο θέμα είναι ότι το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να παράγει ηρωίνη. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να εισάγει τους ε, χημικούς ε, ε, πρόδρομους της ηρωίνης από αυτού πρέπει φυσικά να παρέμβουμε. Να συνεργαστούμε περιφερειακά με τις χώρες που πιθανά θα μπορούσαν να είναι χώρες διέλευσης. Ακόμα και αν σκεφτεί κανείς ότι εισάγονται διάφοροι τόνοι προδρόμων ουσιών, είναι μεγάλες ποσότητες, είναι ορατές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει κάποιο είδους έλεγχος καλύτερος. Εδώ αυτό γίνεται όλο ένα και περισσότερο γνωστό, ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση πιο οργανωμένη στο θέμα. Μια σύντομη αναφορά στο θέμα της εκρίζωσης. Περάσαμε από μια περίοδο όπου η εκρίζωση δεν θεωρείται απαραίτητη. Υπόθηκε επίση ότι ίσως κάποια τμήματα ε, ε, κρίζωση θα έπρεπε να γίνουν, ε, δηλαδή target eradication, έτσι είχε ονομαστεί αυτή η υπόθεση. Για τι αστυνομικέ δυνάμει τώρα. Πιστεύω έχουμε ήδη μία αξιολόγηση για τις αστυνομικέ δυνάμεις. Αυτό το οποίο ήθελα να πω όμως είναι ότι η φαινομενική κατακαιρματισμένη φύση των αστυνομικών δυνάμεων που παρουσιάζεται σε σχέση με την αστυνομία είναι μόνο φαινομενική. Υπάρχει ένα σώμα που λέγεται IPCB που είναι μια τζίργα, δηλαδή μια συνέλευση όπως λένε οι Αφγανοί και συνενώνει, συν, συνέρχονται σε αυτό όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της ε, και συμμετέχουν και οι Αμερικανοί και η UPOL. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία ότι η UPOL, η, ο επικεφαλής της UPOL τουλάχιστον, προεδρεύει αυτή τη ομάδα μέσα στο IPCB <clears throat> που ασχολείται με τις στρατηγικές σε τεχνικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν καλή συνεργασία. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και ακόμα και αν είναι διαφορετική η προσέγγιση μεταξύ αυτών, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε επιτυχώς το πρόβλημα της συνεργασίας και του συντονισμού των διαφόρων προσεγγίσεων. Πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν, αλλά παρόλα αυτά βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Για για την σημαντική <clears throat> πρόοδο. Ποια είναι η πιο σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Κάτι το οποίο θεωρείται πραγματική ιστορία επιτυχίας είναι αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της υγείας. 80% των Αφγανών πολιτών σήμερα καλύπτονται από τις ιατρικές υπηρεσίες. πριν από τρία χρόνια, ίσως ήταν μονάχα 30% που καλυπτόντουσαν από αυτές οι υπηρεσίες. Αυτό είναι μια πραγματική πρόοδος λοιπόν. Αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το οποίο εγώ ονομάζω βασικές υπηρεσίες. Και θα προχώρησε ακόμα περισσότερο αυτό. Ήδη από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε μια εκστρατεία για εμβολιασμό ακόμα και σε περιοχές ε, του, της χώρας όπου υπάρχει ισχυρό ανταρκτικό κίνημα. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό σημαίνει ότι οι βασικές υπηρεσίες και η παροχή βασικών υπηρεσιών όπως είναι χάρη, ο εμβολιασμός σε ευραία στρώματα του πληθυσμού, ιδίως τα πιο τροτά όπως είναι τα παιδιά, ήταν τόσο επιτυχής η πρόθεση αυτών των υπηρεσιών που ακόμα και τα Ταλιμπάν έχουν συνεργαστεί. Επρόκειτο στη συγκεκριμένη περίπτωση για εμβολιασμό κατά της πολιομιελίτιδος. Νομίζω ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι αυτές που δεν έχουν ακόμα έρθει στην επιφάνεια, δεν είναι φανερές και νομίζω είναι στον τομέα της διακυβέρνησης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο η σχέση του ΝΑΤΟ με τη Γιούπολ. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία γιατί σε τοπικό επίπεδο υπάρχει κατανόηση του γεγονότος <clears throat> ότι είτε θα είμαστε μαζί ή αλλιώς θα κάνουμε δύο χωριά. Και το ΝΑΤΟ δίνει διευκολύνσεις στην UPOL και υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο ώστε να υπάρχει χρηματοδότηση μέχρι 80% προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Αποστολή. Αυτό δεν είναι συνεργασία αυστηρά τη ενία με τον ΝΑΤΟ, αλλά είναι μια μορφή συνεργασίας που δείχνει ότι εμεί προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κατακαιρματισμού που χαρακτηρίζουν ακόμα και τη διεθνή παρουσία στο Αφγανιστάν. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, μιλήσατε για τις ευρωπαϊκές φυλές. Πρέπει να σας πω ότι την πρώτη φορά που συνάντησα τον Καζάη, με ρώτησε τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα. και προσπάθησα να το εξηγήσω με τον πιο ευγενικό και σαφή δυνατό τρόπο τι κάνω. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη είναι λιγάκι σαν το Αφγανιστάν. Υπάρχουν πολλές φυλές. Κάθε τόσο κάνουμε μια ζύργα για να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις στις τέντες μας στις Βρυξέλλες. Για μένα, για το Αφγανιστάν, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να φέρουμε από κοινού τις ε, διάφορες φυλές. Αυτό κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και εγώ αυτό κάνω. Το κατάλαβα. Δεύτερος γύρος. Δυστυχώς, ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω. Θα πρέπει να περιοριστεί σε μονόλεπτες παρεμβάσεις, γιατί ο κύριος Πρέπει θα πρέπει να μπορέσει να απαντήσει και να φύγει κιόλας στις 16.45 ε, το αργότερο. Παρακαλώ λοιπόν να μείνετε στο ένα λεπτό και έτσι να μπορέσετε όλοι να μιλήσετε. Ο κύριος Κασουλίδης πρώτα. Thank you, Chairman. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και η Ευρώπη πρέπει να περιμένουν έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το Αφγανιστάν ε, δεν θα προσφέρει καταφύγιο στους ε, τρομοκράτες. Έχουμε λοιπόν ε, περισσότερους θανάτους με την πάρα του χρόνου και οι Αμερικανοί ζητούν να σταλούν ε, περισσότερα στρατεύματα στο Αφγανιστάν. Η εναλλακτική λύση είναι να στηριχθεί η κυβέρνηση. Εσείς ε, ο ίδιος είπατε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να εμπνέει αξιοπιστία και λογοδοσία και δέσμευση. Φοβάμαι λοιπόν ότι η κυβέρνηση η οποία έχει εμπλακεί σε τέτοια κλίμακα σε αμάτες, πώς μπορεί να είναι αξιόπιστη και υπεύθυνη κυβέρνηση. Και εάν υπάρχει ένας ε, δεύτερος ε, γύρος, ε, μήπως ο άλλος υποψήφιος μπορεί να είναι αξιόπιστες. Ο κύριος Τάλερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο να υπάρχει μια στρατηγική θα ήθελα, ε, κύριε Πρέσβη, να γνωρίζω την άποψή σας ε, για το εξής. Κοιτάξτε, η δική μας η στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν, κατά την άποψή σας, δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δεν φοβάστε ότι θα αυξηθεί η βία και ο αριθμός των Ταλιμπάν. Δεν νομίζετε ότι έχει φτάσει πια στιγμή να αποσύρουμε τις στρατιωτικές μας δυνάμεις από το Αφγανιστάν με βάση αυτά που μας ε, είπαν πριν, είπατε πριν από ένα ή δύο χρόνια. Τότε η κατάσταση ήταν καλύτερη. Σήμερα έχει επιδεινωθεί και από το πρίσμα της ασφάλειας και από το πρίσμα της κόπωσης. Έτσι λοιπόν ερωτώ, ποιος είναι ο λόγος ε, που ε, δεν μπορούμε να βρούμε μια στρατηγική για να βελτιωθεί η κατάσταση. Μήπως έχει φτάσει λοιπόν η χρονική στιγμή να βρούμε μια εναλλακτική λύση, να ε, μπορέσουμε στο Αφγανιστάν να ενσωματώσουμε σε μια στρατηγική ότι δεν είναι ακραίο. Και με τον τρόπο αυτό να μην συνεχίσουμε να θρέφουμε την αυταπάτη ότι εμείς τελικά θα αναλάβουμε την διαχείριση αυτή τη χώρα. Ο κύριος Βαν Μπάλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο ε, κατά πόσο εμείς πιστεύουμε ότι οι εκλογές στο Αφγανιστάν ε, ήταν αδιάβλητες και νόμιμες ή όχι. Θα ήθελα να μας πείτε ε, το εξής. Ο πρόεδρος κύριος Καρζάη μέσα στη χώρα του χέρι αξιοπιστίας, ναι ή όχι, με βάση αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν. Λοκ Μπίλερ, επόμενος. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να φερθώ λιγάκι στις ε, εκλογές από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν ακούσαμε ότι έκανε μια σύγκριση με τις εκλογές του 4 και του 5 και διαπιστώθηκε ότι πολλές γυναίκες τώρα ναι μεν μπορούν να ψηφίσουν αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να το πράξουν γιατί είναι απογοητευμένε από τις εξελίξεις. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις. Και ακούσαμε πολλές περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνή κοινότητα πολύ αργά σκέφτηκε να μπορούν οι γυναίκες να πηγαίνουν σε εκλογές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, ε, σίγουρα το έχετε ακούσει και εσείς αυτό, ερωτώ ε, Τώρα πλέον, τι είδου ε, μάθημα έβγαλε κανεί, ε, θα είναι οι γυναίκε περισσότερο προστατευμένε και περισσότερο ενημερωμένε όταν την επόμενη φορά θα κληθούν να ψηφίσουν για τι προεδρικέ εκλογέ. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν για ένα λεπτό. Ναι, πρόεδρε. Ε, πολύ μεγάλο σεβασμό έχω και μεγάλη τιμή στο πρόσωπο του ε, πρέσβεως, ε, του Ξέρετε ότι όλο και λιγότερο ο ευρωπαϊκός πληθυσμός θέλει να συμμετέχουν ε, οι ευρωπαϊκές χώρες εκεί. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε και την κατάσταση έτσι για να αλωνίζουν. Εσείς όμως πώς το βλέπετε αυτό και πώς το συζητάτε με τους ενδιαφερομένους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βόμποντα, ένα λεπτό. Κοιτάξτε, εγώ έχω μόνο μία ερώτηση να κάνω. το να κάνει κανείς ε, τη δουλειά του, όπως την κάνετε εσείς και όπως την κάνουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πόσο καιρό θα είναι απαραίτητη ισχυρή στρατιωτική παρουσία. Μιλήσατε για κόκκινες γραμμές, συμφωνώ. Αλλά εσείς για πόσο καιρό πιστεύετε ακόμα θα χρειαστεί ε, στρατιωτική παρουσία. Δύο, πέντε, δέκα χρόνια πόσα. Αυτό θα με ενδιαφέρε. Ευχαριστούμε Κύριε Σβόμποντα, το λόγο η κυρία Σάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταλαβαίνω πολύ καλά τις ε, δυσκολίες που έχετε σχετικά με τις φυλές και εδώ και στο Αφγανιστάν. Μιλήσατε για την αναξιοπιστία των θεσμών και θέλω να ρωτήσω κατά πόσον τα στατεύματά μας ε, έχουν συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση που βεβαίως ε, σίγουρα έχουν τις καλύτερες των προθέσεων αλλά υπάρχουν κάποιες υπόνοιες ε, για τις οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζονται οι δικές μας οι ευρωπαϊκές. Αυτές κατηγορούνται για αδικίες, για απάτες, και θέλω να γνωρίζω ε, τι είδους ε, μηχανισμούς ασφαλείας έχετε. Γιατί οι δικοί μας άνθρωποι εκεί είναι για να βοηθήσουν τους Αφγανούς και όχι για να κατηγορούνται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απάτες. Λούνα Τσεκ, ε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σέκη, εσείς είπατε ότι εναπόκειται στους Αφγανούς να αποφασίσουν για το ποιον θέλουν να έχουν πρόεδρο. Πρόσφατα όμως ακούσαμε ότι υπήρξε μια διάσπαση. Ε, ο κ. Κάλπρεϊθ αναγκάστηκε να φύγει ε, γιατί δεν υπήρχε σύνδεση απόψεων για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Υπάρχουν υπόνοιες ε, μεγάλων απατών και ανησυχώ πάρα πολύ για το ότι και εσείς και τα Ηνωμένα Έθνη κατά κάποιον τρόπο τα απορρίπτεται όλα αυτά και λέτε εμείς θα συνεχίσουμε τον Καρζάη ό,τι και αν έγινε. Εάν λοιπόν πιστεύετε ότι ε, εναπόκειται στους Αφγανούς να αποφασίσουν, θα πρέπει να δείτε και αυτές τις υπόνοιες. Και όχι να συνεχίσετε να ε, συνεργάζεστε με τον ε, Καρζάη, να μην έγινε τίποτα. Τι λέτε από αυτού για τις υπόνοιες της απάτης. δεν νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος που προσεγγίζει το θέμα, ότι ο τρόπος που προσεγγίζει το θέμα είναι και ο καλύτερος. Ο αντιπρόεδρος Πασκού γιατί για 1,5 λεπτό, επειδή είναι αντιπρόεδρο, δίνουμε και 30 δευτερόλεπτα παραπάνω. Κοιτάξτε, και εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ε, παρουσίασή σας. Εγώ έχω την εντύπωση ότι όσο πιο πολύ μείνουμε, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Αν πάτε παραδείγματο χάρη την θέση των Ταλιμπάν το 2001, το 2 και τη συγκρίνετε με τη θέση τους τώρα, θα διαπιστώσετε ότι οι Ταλιμπάν επανήλθαν και μόνον αυτό αλλά μας ε, έχουν φέρει σε πολύ δυσχερέστερη κατάσταση από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Πόσο λάβαμε υπόψη μας την παράδοση στο Αφγανιστάν, σε αυτό που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ως ε, κράτος, ε, θεσμούς, αστυνομία, οτιδήποτε το οποίο πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κράτος για να μην ξαναγίνει το Αφγανιστάν ε, ένα προπύργιο των τρομοκρατών. Σας ευχαριστώ. Παρά ότι σας έδωσα μπόνους 30 δευτερόλεπτα, <laughs> μιλήσατε λιγότερο από ένα λεπτό. Έχουμε απλά το χρόνο για να απαντήσετε 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πριν να απαντήσω, κάτι το οποίο ξέχασα να σας πω προηγουμένως το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Με ρώτησε κάποιος βουλευτής πώς συνδυάζουμε τη συμφιλίωση με τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών. Θα σας αφηγηθώ μια ιστορία η οποία νομίζω ότι έχει πραγματικά νόημα. Μου εξηγήσαν με τον πιο σαφή δυνατό τρόπο ποια είναι η κατάσταση μου το είπε μια βουλευτής του Μπαϊάμ, της περιοχής του Μπαμπιάμ, του τοπικού συμβουλίου. Μου είπε ότι αν συμφιλίωση σημαίνει να μην είμαι πια μέλος αυτού του συμβουλίου, να μην μπορώ να είμαι υποψήφια για ένα δημόσιο αξίωμα, να μην πηγαίνουν τα κορίτσια στο σχολείο, ξεχάστε το. Αν μπορώ να συνεχίσω να δρώ στην πολιτική ζωή, το συζητάμε. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή την οποία ήθελα να υπογραμμίσω. Και θα ήθελα <clears throat> να αντιμετωπίσω το θέμα των... της απάτης συνολικά. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση της Νοθείας στο Αφγανιστάν. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα θέματα αυτά και η εντολή μου αναφέρει σαφώς ότι μεταξύ άλλων εγώ πρέπει να υποστηρίξω την δημοκρατική αυτή διαδικασία. Προσπαθώ να το κάνω με, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι μια λυπηρή ιστορία. Γιατί έχω προσωπική φιλία και με τον Πίτερ Κάμβιατ και με τον Καγιάε Να το θέσω διαφορετικά το θέμα είναι φανερό ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε νοθεία και ατασταλίες. Αν με ρωτήσετε αν υπήρξαν ατασταλίες και ανομαλίες, ναι, η απάντηση είναι ναι. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η έκταση αυτών των ατασταλιών, δεν ξέρω, η απάντησή μου. Και περιμένω από τους αρμόδιους θεσμούς, οι οποίοι πρέπει να ελέγξουν την εκλογική διαδικασία, και ιδίως την εκλογική επιτροπή για τα παράπονα που αποτελείται από πέντε μέλη τρία εκ των οποίων δεν είναι Αφγανοί να ερευνήσουν όλες αυτές τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί. Τότε θα μπορούσα να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα όταν περατωθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω σίγουρα είναι να πω ότι εγώ υποστηρίζω μια διαδικασία η οποία, όπως είπα και στην αρχή, βασίζεται στην εκλογική Επιτροπή Παραπώνων και την Ανεξάρτητη Επιτροπή Παραπώνων. Δεν θέλω λοιπόν να δυσκολεύσω το έργο τους με το να υπονομεύσω ήδη από την αρχή το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όποιο και να το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για την αξιοπιστία <clears throat> του Πρόεδρου, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρίνουν οι ίδιοι Αφγανοί και ο πιο εύγλωτος τρόπος για να το πράξουν είναι με τις ψήφους τους. Και η Επιτροπή για τα εκλογικά για τα παράπονα σε σχέση με την πληροφορία θα ελέγξει όλες τις καταγγελίες. Ο ρόλος των γυναικών ο ρόλος των γυναικών στην πολιτική στο Αφγανιστάν. Είναι ένα σημαντικότατο θέμα. Οι γυναίκες κοινοβουλευτικοί στο Αφγανιστάν θα έλεγα και το λέω με απόλυτη επίγνωση της ευθύνης που έχω είναι πολύ καλύτερες από τους άρενες συναδέλφους τους. Και αυτή είναι μια άποψη που δεν την έχω μόνο εγώ, τη συμμερίζονται πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι η προσέλευση στις κάλπες, από ό,τι βλέπουμε από τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε, η προσέλευση των γυναικών ήταν περιορισμένη. Τα καλά νέα όμως είναι ότι ο αριθμός των εκπροσώπων, των γυναικών εκπροσώπων που εξελέγησαν στα περιφερειακά συμβούλια, είναι υψηλότερος από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές. Και αυτά είναι θετικά. Γιατί στο τοπικό επίπεδο υπάρχουν πολλές, ας το πω έτσι, πιέσεις τις οποίες γνωρίζουμε. Πώς μπορούμε τώρα να ενισχύσουμε το ρόλο των γυναικών στις, επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές. Το είπα προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι μια γενική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας. Είναι μια ευθύνη και των αφγανικών θεσμών, αλλά είναι και ευθύνη των κοινοβουλευτικών από άλλες χώρες. Ο λόγος για τον οποίο έχω κάνει μια έκκληση προς εσάς να είστε περισσότερο παρόντες στην διαδικασία την εκλογική του, του Αφγανιστάν ακόμα και πριν από τις εκλογές είναι ακριβώς για να ενισχύσετε πάνω απ' όλα αυτές τις γυναίκες οι οποίες είναι ιδιαίτερα θαραλέες και αγωνίζονται για τη δημοκρατία και οι οποίες μπορούν να δώσουν μια μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της δημοκρατίας στη χώρα τους. Και θα έλεγα ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή τη χώρα θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στην διατήρηση της σταθερότητας του Αφγανιστάν για πολύ καιρό. Τώρα το θέμα τι θέλετε, το θέμα της στρατιωτικής μας παρουσίας. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί. Πού να ξέρω. Δεν είμαι στρατηγός, δεν είμαι σε θέση να προβλέψω το μέλλον. Αυτό το οποίο λέω είναι διαφορετικό. Ότι χρειάζεται να επιταχύνουμε τη διαδικασία της μεταβίβασης τους Αφγανούς, στους Σύριους, της εξασφάλισης της ε, ασφάλειας. Η λεγόμενη αφγανοποίηση. Αυτό είναι λοιπόν προϋπόθεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Για τη Νοθεία νομίζω ότι απάντησα ήδη. Οι αφγανικές παραδόσεις. Έχετε δίκιο, αυτό είναι σημαντικό θέμα. Πού βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ των αξιών της αφγανικής κοινωνίας και των δημοκρατικών αξιών που προωθούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους στόχους της διαδικασίας αφγανοποίησης. Εγώ πέρασα πέντε χρόνια στο Αφγανιστάν. Η εμπειρία μου και η εντύπωση που έχω είναι ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη υπερηφάνεια σε όλα τα επίπεδα των Αφγανών που μπορούν να ελέγχουν όλο και περισσότερο την τύχη τους και να έχουν τα ενία της χώρας τους. όχι μονάχα έναντι των ξένων, των δυτικών. Να σας πω μια ιστορία. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι ε, διοικητής μιας περιοχής στο ανατολικό μέρος του Αφγανιστάν, στο Κουμάρ. Έρχεται μια μέρα να με δει αυτός ο διοικητής, ο οποίος με είχε βοηθήσει πάρα πολύ το 2005 όταν είχα να αντιμετωπίσω την απαγωγή μιας Ιταλίδας. Εγώ χρησιμοποιώ λοιπόν αυτή την ευκαιρία της παρουσίας του για να ακούσω την άποψή του. Τελευταία φορά που τον, τον συνάντησα, τον ρώτησα τι πιστεύεις για την ε, συμφιλίωση, εθνική συμφιλίωση. Μου λέει πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ Αφγανών Ταλιμπάν και ξένων Ταλιμπάν. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί ξένοι Ταλιμπάν που έρχονται από άλλες χώρες, από την άλλη πλευρά των σύνορων. Και δεν τους θέλουμε άλλο. Δεν θέλουμε να συνεχίσουν να βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Πιστεύω λοιπόν ότι οι Αφγανοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ποια είναι η δυνατότητα που έχουν ενώπιόν τους και η δυναμική και ξέρουν ότι ποια είναι καιρός να αρχίσουν να ελέγχουν τη χώρα τους. Eh, Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Πραγματικά ήταν ε, πολύ πλούσια και εις βάθος η συζήτηση, παρά τη συντομία που χρειάστηκε να τηρήσουμε και να ευχαριστήσουμε την ευκαιρία του συναδέλφους, αλλά και τον πρέσβη που μπόρεσε τόσο σύντομα να δώσει απαντήσεις σε τόσο περίπλοκες ε, ερωτήσεις ε, και πολύ άριθμες ερωτήσεις. Όπως θυμήσατε και στην αρχή της παρέμβασής σας, ε, ο ευχή ξεκινά σήμερα μια συνεργασία μαζί σας ε, με την Επιτροπή μας, που σίγουρα θα σημάνει και περαιτέρω επαφές. ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε κι εμείς γιατί σε αυτή τη τόσο ταλαιπωρημένη περιοχή του κόσμου να μπορέσουμε να, να, να επικρατήσει η ειρήνη και η δημοκρατία και η ευημερία και η δυνατότητα να ζήσουν επιτέλους όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε μια ε, κανονική και ήρεμη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ε, τέλος της ε, συνεδρίασης αυτής ξαναρχίζει η συνεδρίαση για τον ορισμό των υποψηφίων για το βραβείο Ζαχάροφ, να δώσουμε το χρόνο στους συναδέλφους από την Επιτροπή Ανάπτυξης να έρθουν εδώ στις 5 και 4. Θα τα ξαναλέμε και κλεισμένο το θυρών.